Good morning. Good morning, dear colleagues, dear friends. Please be seated. get started early in the morning. Ας ξεκινήσουμε, είναι νωρίς το πρωί. Είναι από τις τελευταίες μας συνεδριάσεις. Συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελευθεριών των Πολιτών σε αυτήν την κοινοβουλευτική θητεία. Οπότε, ας περάσουμε απευθείας στην έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Δηλαδή, θα προτείνω τις εξής αλλαγές. Σημείο 13α, νέο σημείο στην ημερήσια διάταξη, δηλαδή από τις 12, από τις 12 12.30 θα έχουμε παρουσίαση από την νομική υπηρεσία του Ευρωκοινοβουλίου και της Προεδρίας του Συμβουλίου για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την κράτηση, την τήρηση δεδομένων. Αντιρρήσεις, κάνουμε αυτή την αλλαγή, μετά ανακοινώσεις προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Να σας ευχαριστήσω όλους και πάλι για την σκληρή σας δουλειά και τη συνεργασία που είχαμε και πραγματικά λυπούμε που δεν είναι η καταλληλότερη χρονική στιγμή για να για να συνεχίσουν τη δουλειά μας, αυτοί που θα ακολουθήσουν εδώ, καθώς είναι η επόμενοι, δεν έχει λάβει καθήκοντα η επόμενη Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, αλλά είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε χθες το βράδυ και να αποχαιρετιστούμε. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι όπως ζητήθηκε από τους συντονιστές, η Επίτροπος Μάστρομ ε, έλαβε επιστολή, έστειλε μάλλον η ίδια μια επιστολή χθες, για τα αρχεία τα προηγμένα αρχεία τήρησης δεδομένων για επιβάτες με την, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία της Ρωσίας οι οποίοι θέλουν να εγκαθιδρύσουν ένα σύστημα PNR ε, για όλες τις διεθνείς πτήσεις που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ γύρονται πάρα πολλά ερωτήματα, τέθηκαν πολλά ερωτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά την νομική ασφάλεια μιας τέτοιας διευθέτησης και στο παρελθόν η Επίτροπος μας είχε πει ότι οι ρωσικές αρχές είχαν ε, παράσχεται σχετικέ διαβεβαιώσει ώστε να μην ε, εισάγουν, να μην προβλέψουν τέτοιο σύστημα μονομερό. Ωστόσο, τώρα έχουν προκύψει νέε ανησυχίε, νέοι ενδιασμοί και νέε πληροφορίε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διευκρινήσει για το όλο ζήτημα. Οπότε θα έχουμε ειδήσει από την από την Επίτροπο Μάλστρομ ως προς το τι στοιχεία συγκέντρωσε και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 we are approving the minutes of the last meetings that you got them. I hope there is no objections as to the minutes. Δεν νομίζω να υπάρχουν αντιρρήσεις και θα γνωρίζετε ότι τα πρακτικά της 14ης Νοεμβρίου έχουν μια συγκεκριμένη μνήμα που καλό είναι να σημειωθεί και μια προσθήκη επίσης στην συνεδρίαση της 20 Μαρτίου στα πρακτικά της συνεδρίασης εκείνης. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, περνάμε στο πρώτο σημείο τη συζήτησή μα, την ημερήσια διάταξη, το σημείο 4. Κατάλογο τρίτων χωρών, οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρηση για τη διέλευση των εξωτερικών σύνορων των κρατών μελών. Και κατάλογο των τρίτων χωρών, οι οποίοι εξαιρούνται. Οι οποίε εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή. Έχουμε ψηφίσει την έκθεση Γκάμπριελ στην Ολομέλεια σχετικά. Πριν οι νομομαθείς Οι γλωσσομαθείς νομικοί ε, αποσαφηνίσουν το κείμενο. Οπότε θεωρούμε ότι εγκρίνεται. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Αυτό νομίζω ότι δεν χρειάζεται περαιτέρω συζήτηση. Σημείο 5. Απλουστευμένος έλεγχος προσώπων στα εξωτερικά σύνορα. Και πάλι έγκριση διορθωτικού. Βασιζόμενος στον ε, κανόνα 116. Τον περασμένο Φεβρουάριο, στην ε, τελευταία Ολομέλεια, το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση την πρόταση απόφαση για την εισαγωγή μια απλουστευμένη διαδικασία για τον έλεγχο των προσώπων στα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει και ένα διορθωτικό και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, θεωρούμε ότι εγκρίνεται και αυτό. Και τώρα περνάμε σε μια κοινή συζήτηση επί, επί των σημείων 6, 7 και 8. Θεωρήσεις είναι το βασικό θέμα. Κανονισμός για, την, ε, για τις θεωρήσεις, για τον κώδικα θεωρήσεων και έκθεση προς το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο μια πιο ευθύς πολιτική θεωρήσεων με στόχο την οικονομική ανάπτυξη. Θα έχουμε εδώ παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα παρουσιαστεί έκθεση αξιολόγηση του ισχύοντος ε, κώδικα θεωρήσεων, όπως ισχύει, καθώς και θα δούμε αν θα υπάρξει μια ομοθετική πρόταση για την διόρθωση του ε, κώδικα θεωρήσεων με μια αναδιατύπωση και μια πρόταση για τις λεγόμενες τόρινγκ, ε, τις χειριστικές θεωρήσεις. Για τις ταξιδιωτικές λοιπόν θεωρήσεις που θα υπάρξει ειδικό νομοθέτημα. Τώρα, για την παρουσίαση αυτού του πακέτου, έχετε το λόγο κύριε Ντεκουέστορ. Um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, είναι μεγάλη χαρά και τιμή να είμαι εδώ σήμερα ενώπιον σα για να παρουσιάσω ενώπιον τη Επιτροπή σα το πακέτο για τη μεταρρύθμιση του κώδικα για τη χορήγηση προξενικών θεωρήσεων. Αυτό εγκρίθηκε από την Κομισιόν την προηγούμενη εβδομάδα και για να είμαι πιο συγκεκριμένο, ενεκρίθη την 1η Απριλίου. Δεν ξέρω αν σα λέει αυτό κάτι. Η 1η Απριλίου συνδέεται με τις φάρσες και τα διαφραστία, αλλά δεν επρόκειτο για μια φάση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε μια απόφαση που ήταν το αποτέλεσμα μιας ενδελεχούς ανάλυσης της εφαρμογής του κώδικα προξενικών θεωρήσεων από τα κράτη-μέλη και υπάρχει ένα έγγραφο των υπηρεσιών της Κομισιόν που περιέχει όλες τις λεπτομέρειες του, της εφαρμογής των διαφόρων προνοιών του κώδικα προξενικών θεωρήσεων και τα συμπεράσματα αναφέρονται και στην ε, ανακοίνωσή μας για μια ευφιέστερη πολιτική προξενικών θεωρήσεων. Υπήρξαν και τα αποτελέσματα μιας δημόσιας διαβούλευσης που διοργάνωσε η Κομισιόν. Και όπως ξέρετε, η Κομισιόν θα ήταν υποχρεωμένη να παρουσιάσει μια αξιολόγηση εφαρμογής του κώδικα αυτού τρία χρόνια Και η Κομισιόν δεν περιορίστηκε μονάχα στο να παρουσιάσει αυτή την έκθεση, αλλά συγχρόνως ενέκρινε και δύο νομοθετικές προτάσεις. Η μία για να υπάρξει ε, τροποποίηση και αναμόρφωση του κώδικα για τις θεωρήσεις και μια δεύτερη απόφαση νομοθετικού χαρακτήρα για τη δημιουργία της λεγόμενης τουριστικής ή ταξιδιωτική βίζας. Στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Φεβρουάριο είχαν διατυπωθεί κάποιες ε, επικρίσεις σε σχέση με την προξενική θεωρήσεων και γι' αυτό η Κομισιόν θεώρησε σκόπιμο να έρθει με νομοθετικές προτάσεις. Μάλλον υπήρξε επικρίση γιατί η Κομισιόν ήρθε αμέσω με νομοθετικέ προτάσει. Το Κοινοβούλιο θεώρησε ότι πρώτα η Κομισιόν θα πρέπει να κάνει μια αξιολόγηση, να κάνει διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα και μετά να προχωρήσει στην κατάθεση νομοθετικών προτάσεων. Σε σχέση με το θέμα αυτό όμω, κύριε Πρόεδρε, θέλω να αναφέρω ότι ήδη στην ανακοίνωσή της στη Κομισιόν για τη συμμετοχή των προξενικών θεωρήσεων στην οικονομική ανάπτυξη, η Κομισιόν ανέφερε μια πληθώρα προβλημάτων που αντιμετωπίζαμε με την εφαρμογή του κώδικα για τις θεωρήσεις. Για να επιταχυνθεί λοιπόν η διαδικασία αυτή και να θεραπευθούν τα προβλήματα τα οποία είχαν διαπιστωθεί, η Κομισιόν αποφάσισε να συνοδεύσει την πολιτική αυτή έκθεση με τις νομοθετικές προτάσεις που έχετε ενώπιόν σας. Με τον τρόπο αυτό θεωρούσε ότι θα μπορέσει να διευκολύνει τη συζήτηση και να επιταχύνει, ελπίζουμε, την έγκριση νέων μέτρων στον τομέα αυτό. Ήδη έχω αναφέρει τις δυσκολίες που υπήρξαν στην εφαρμογή του κώδικα θεωρήσεων. Ήταν όλα αυτά τόσο τραγικά? Όχι, θα έλεγα. Αν δείτε τα στοιχεία του 2013, πάνω από 17 εκατομμύρια αιτήσει για βίζα στον χώρο του Σέγγεν είχαν υποβληθεί. Ενώ το 2009, σε σχέση μάλλον με το 2009, υπήρξε μια αύξηση 68,5% για αιτήσει βίζων προξενικών θεωρήσεων Σέγγεν. Είναι μια επιτυχία λοιπόν. Υπάρχουν όμως πολλές δυνατότητες. Τα 17 εκατομμύρια είναι ένας εντυπωσιακός αριθμός αλλά έχουμε και άλλα εντυπωσιακά ε, αριθμητικά στοιχεία. Εκτιμάται ότι τουλάχιστον 6,6 εκατομμύρια δυνητικοί επισκέπτες δεν μπήκανε στην περιοχή του Σέγγεν το 2011 λόγω του επαχθούς καθεστώτος και της ε, μεγάλης γραφειοκρατίας που απαιτεί το. Αυτές οι εκτιμήσεις είναι κάτι που πρέπει να δώσει λαβή σε ενέργειες από την Κομισιόν. Κάθε χρόνο πολλοί δυνητικοί τουρίστες αποθαρρύνονται από το να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι μόνο ένα πρόβλημα για αυτούς που θέλουν να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σημαντική οικονομική απώλεια για την ευρωπαϊκή οικονομία. Δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε τα ωφέλη που θα μπορούσαν να προκύψουν από αυτούς τους τουρίστες. Και για να συνεχίσω με στοιχεία, η διευκόλυνση της διαδικασίας προξενικών θεωρήσεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση ταξιδιών προς τη ζώνη του Σέγγεν κατά 60%. Μέσα σε πέντε χρόνια αυτό θα σήμαινε 130 δισεκατομμύρια σε άμεσες δαπάνες για στέγαση, μεταφορές, ψυχαγωγία και αγορές. Περίπου 1,3 πρόσθετε θέσει εργασία στον τουρισμό θα μπορούσαν να προκύψουν από μια τέτοια διευκόλυνση. Για να μπορέσουμε λοιπόν να αποκομίσουμε αυτά τα ωφέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να έχει μια πιο ευφυή και κοινή πολιτική για τι προξενικέ θεωρήσει. Μπορούμε να ενισχύσουμε τη δημιουργία θέσεων απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη με το να έχουμε μια πιο οικονομική διάσταση στην πολιτική μα για τι θεωρήσει, ενώ συγχρόνω θεωρούμε να εξασφαλίσουμε το υψηλότερο επίπεδο ασφάλεια στα σύνορά μα. Και εδώ αναφέρομαι στην εκθέση τη κυρία Γκάμπριελ, η οποία επιβεβαιώθηκε από εσά σήμερα το πρωί, μέσα στα κριτήρια που αναφέρει για τη θέσπιση του καταλόγου προξενικών θεωρήσεων, έχει προσθεθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το οικονομικό όφελος και τα ωφέλη που έχουν να κάνουν με το εμπόριο και τον τουρισμό και αυτό είναι ένα από τα κριτήρια που, λαμβάνουμε, που θα λαμβάνουμε υπόψη όταν αναθεωρούμε τους καταλόγους για τις προξενικές θεωρήσεις. Αυτό είναι και μια διάσταση που η Κομισιόν έλαβε υπόψη της στα πλαίσια της αξιολόγησης εφαρμογής του κώδικα για τις θεωρήσεις και όταν εξετάζει ε, βελτιώσεις που θα μπορούσαν να επέλθουν σε αυτόν τον κώδικα. Σας είπα ότι υπάρχουν δύο νομοθετικές προτάσεις. Η πρώτη είναι μια τροπολογία και ε, αναδιατύπωση του κώδικα για τις προξενικές θεωρήσεις. Ο κώδικας αυτός έφερε σημαντικές βελτιώσεις έναντι της κατάστασης που υπήρχε στο κεκτημένο, το διακυβερνητικού χαρακτήρα κεκτημένο του Σέγγεν για τις θεωρήσεις. Ήταν μια πρώτη επανάσταση αν θέλετε. Πιστεύουμε όμως ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε και σε μια δεύτερη επανάσταση ώστε να επιφέρουμε σημαντικές βελτιώσεις στον κώδικα αυτό. Είναι σαφές ότι πολλοί ετούντες θεωρούν ότι είναι πολύ μακροσκελής και πολυδάπανες οι διαδικασίες. Χρειάζεται πολύς χρόνος σε ορισμένα προξενικά γραφεία για να πάρει κανείς ένα ραντεβού. Υπάρχουν καθυστερήσεις για την έκδοση της βίζας. Πολύπλοκοι κανόνες σε σχέση με τα συνοδευτικά έγγραφα και διαφορετικές πρακτικές μεταξύ κρατών μελών στις προξενικές αρχές τους. Γι' αυτό η Κομισιόν πιστεύει ότι θα πρέπει να βραχύνουμε τη διαδικασία <clears throat> αίτησης, για παράδειγμα ο χρόνος επεξεργασίας των αιτήσεων αυτών δεν θα πρέπει να ξεπερνάει 10 ημερολογιακές μέρες, ενώ σήμερα είναι 15 μέρες βάσει του κώδικα θεωρήσεων. Θα πρέπει να απλοποιήσουμε επίσης τους κανόνες σε ό,τι αφορά τα συνοδευτικά έγγραφα. Θα πρέπει εξάλλου να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη εναρμόνιση για τον κατάλογο των συνοδευτικών εγγράφων που ζητούν τα προξενία των κρατών μελών για κάθε τουριστική βίζα. Η πρότασή μας επίσης αναφέρει με σαφήνεια ότι ορισμένε κατηγορίες ετούντων μπορούν να κάνουν την αίτησή τους στο διαδίκτυο επιγραμμικά. Και υπάρχει και μια επέκταση των κατηγοριών που δεν, των ετούντων που δεν χρειάζεται να πληρώσουν τέλη για την απόκτηση προξενικής θεώρησης. Έχουμε πολλά παράπονα εξάλλου από αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να <clears throat> υποβάλουν την αίτησή τους στην χώρα όπου διαμένουν. Γιατί τα κράτη-μέλη εκεί δεν έχουν προξενικές αρχές ή δεν εκπροσωπούνται σε προξενικό επίπεδο στη χώρα αυτή. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί και να βελτιωθεί ώστε να εξασφαλιστεί ότι ένας ετών μπορεί πάντα εκεί που μένει να κάνει μια αίτηση για προξενική θεώρηση. Γι' αυτό η Κομισιόν στην πρότασή της προβλέπει ένα σύστημα υποχρεωτικής εκπροσώψης που υποχρεώνει τις ε, παρούσες εκεί προξενικές αρχές να δεχτούν αιτήσει για άλλα κράτη-μέλη τα οποία δεν εκπροσωπούνται ή δεν είναι παρόντα. Λίγη ακόμα λεπτομέρεια για το θέμα αυτό. Ορισμένοι ετούντες πρέπει να ταξιδέψουν και να πάνε σε μια γειτονική χώρα για να κάνουν την αίτηση για βίζα, για να μπουν στη ζώνη του Σέγγεν. Στις χειρότερες περιπτώσεις πρέπει πρώτα να ζητήσουν μια βίζα για να πάνε στη χώρα όπου υπάρχει το προξενείο, ώστε να μπορέσουν να πάνε εκεί και να κάνουν την αίτηση για να μπουν στη ζώνη του Σέγγεν. Αυτό είναι μια κατάσταση που σίγουρα δεν θα πρέπει να την ε, διατηρήσουμε. Μία, ένας από τους ακρογωνίες λίτους της ε, αναδιατύπωσης του κώδικα αυτού είναι κάτι που πιστεύει η Κομισιόν ότι θα πρέπει να εισαχθεί στη διαδικασία αυτή με διάκριση από τη μία πλευρά μεταξύ αυτών που δεν είναι γνωστοί στα προξενία της ζώνης του Σέγγεν, δεν έχουν ιστορικό σε σχέση με προξενικές θεωρίες αυτού του είδους και για τους οποίους θα πρέπει να συνεχίσουν καταρχήν να εφαρμόζονται οι τρέχοντες κανόνες αλλά και για αυτούς θα μπορούσαν να υπάρχουν κάποιες διευκολύνσεις σε σχέση με το τωρινό σύστημα και μετά έχουμε την κατηγορία των τακτικών ταξιδιωτών που βρίσκονται στο σύστημα καταγραφής προξενικών θεωρήσεων και έχουν ένα ιστορικό, ένα σαφές ιστορικό για προξενικές θεωρήσεις μέσα στο Σέγγεν. Για αυτού, η Κομισιόν πιστεύει θα πρέπει να περιορίσουμε τη διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών σε σχέση με την ε, διάρκεια ε, ζωή μιας βίζας πολλαπλών εισόδων και να υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια τα οποία εάν εκπληρούνται, αν η προηγούμενη βίζα που έχει πάρει το ενδιαφερόμενο άτομο έχει ληφθεί με σύνομο τρόπο, τότε θα πρέπει να εκδοθεί μια βίζα πολλαπλών εισόδων με διάρκεια τριών ετών. Και αν χρησιμοποιηθεί σωστά και νομίμως αυτή η βίζα, τότε το ενδιαφερόμενο άτομο θα πρέπει να πάρει μια βίζα πολλαπλών εισόδων πενταετούς διάρκειας. Αυτό είναι λοιπόν μια διευκόλυνση που προβλέπει η πρόταση της Κομισιόν ήδη σήμερα τα κάτι μέρη. Έχουν τη δυνατότητα να δώσουν σε ταξιδιώτες καλή πίστη μια βίζα που να έχει διάρκεια μέχρι πέντε έτη, αλλά στην πράξη αυτό είναι η εξαίρεση της εξαίρεσης. Πιστεύω όμως ότι αυτό θα αποτελέσει μια σημαντική βελτίωση η οποία προβλέπεται στην πρόταση της Κομισιόν. Άλλο ένα θέμα τώρα. Και φυσικά δεν μπορώ να τα πω όλα διότι δεν θα μείνει χρόνο στην Επιτροπή σα. Είναι πάρα πολλά στοιχεία που, είναι η, που έχει πρόταση η Κομισιόν είναι η διευκόλυνση των οικογενειακού χαρακτήρα επισκέψεων για μέλη οικογενειών πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν καλύπτονται από την οδηγία του 2004 για την ελεύθερη κυκλοφορία πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των μελών των οικογενειών των. Η οδηγία αυτή επιβάλλει να υπάρχουν διευκολύνσεις όταν αυτά τα μέλη οικογενειών πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση ζητούν μία βίζα, αλλά πολλέ οικογενειακε επισκεψει δεν καλύπτονται από αυτή την οδηγία. Παραδείγματο χάρη, τα μέλη μια οικογένεια ενο πολίτη που έρχονται να επισκεφθούν κάποιον ο οποίος ζει σε μια χώρα μέλος όπου έχει, έχει την, εθνικο, την υπηκότητά του. Σήμερα δεν έχουν καμία ιδιαίτερη διευκόλυνση, απλώς υπόκειται στο γενικό πλαίσιο του κώδικα θεωρήσεων. Αυτά λοιπόν εν γέννη και συνοπτικά είναι οι βασικές αλλαγές που προέρχονται από την αναδιατύπωση της, ε, του, κώδικα θεωρήσεων. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία για την προξενική οργάνωση, αλλά δεν πρόκειται να σας καταπονήσω με τις λεπτομέρειες. Κάτι ακόμα για την πρόταση για την τουριστική βίζα. Από την πλευρά της Κομισιόν έχουμε προετοιμάσει μια χωριστή πρόταση, γιατί αυτή η πρόταση δεν εφαρμόζεται μονάχα σε ανθρώπους που χρειάζονται βίζες για σύντομη ε, παρουσία και παραμονή, αλλά και για αυτούς οι οποίοι έρχονται από τρίτες χώρες που, όπου ισχύει εξαίρεση από τις προξενικές θεωρίες. Όταν αντιμετωπίζαμε τη μεταρρύθμιση του προξενικού κώδικα, Είδαμε ότι είχαμε πολλά παράπονα για το γεγονό ότι υπάρχει ένα νομικό κενό στην νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση για άτομα τα οποία θέλουν να ταξιδέψουν στην περιοχή του Σέγγεν και να σε σερβιανίσουν για διαστήματα από 90 μέχρι 180 ημέρες, όπως λέει ο ορισμός για τη σύντομη παρουσία. Πολλές φορές είναι καλλιτέχνες όπως το ε, που θέλουν να πάνε παραγωγικά να μείνουν ένα μήνα στην Ισπανία, ένα μήνα στην Γαλλία, δύο μήνες στη Γερμανία όμως τελικά μπορεί να φτάσουν σε ένα τουρ το οποίο θα καλύψει ένα χρόνο, ένα μισή χρόνο. Αλλά δεν υπάρχει κανένα σύστημα, δεν υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο που να τους επιτρέψει να κυκλοφορούν στην περιοχή του Σέγγερ για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Πέραν πάσης αμφιβολίας. Υπάρχουν τουρίστες, υπάρχουν καλλιτέχνες, υπάρχουν ερευνητές που έχουν θεμητό συμφέρον να μπορούν να κυκλοφορούν στην περιοχή του Σέγγεν για περισσότερο από 90 ή 180 ημέρες. Γι' αυτό το λόγο εμείς ως Κομισιόν έχουμε προετοιμάσει μια δεύτερη πρόταση διότι και αυτή ανταποκρίνεται στις ανάγκες ορισμένων κατηγοριών ταξιδιωτών και θα αποφέρει οικονομικά ωφέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω κύριε Πρόεδρε ότι με τις προτάσει αυτέ η Κομισιόν προτείνει να προχωρήσουμε σε μια δεύτερη επανάσταση στον τομέα της πολιτικής προξενικών θεωρήσεων. Ελπίζω ότι οι συνομοθέτε θα ακολουθήσουν στην κατεύθυνση αυτή. Υπάρχουν πολλέ καινοτομίε, βέβαια. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων συμφερόντων και συγκεκριμένα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί σωστά η περιοχή του Σέγγεν και δεν θα θυγεί αυτή η λειτουργία γιατί τα οικονομικά ωφέλη πηγαίνουν προς μια κατεύθυνση αλλά συγχρόνω πρέπει να επανεξισορροπηθούν έναντι της ανάγκης ασφάλειας στην περιοχή του Σέγγεν ώστε να μπορέσει να διατηρηθεί αυτός ο χώρος χωρίς εσωτερικά σύνορα να λειτουργεί ευθέτως. Αυτά λοιπόν κύριε Πρόεδρε, αυτά συνοπτικότατα, πάρα πολύ συνοπτικά, είναι τα στοιχεία για το πακέτο μεταρρύθμισης του τελωνιακού, του κώδικα μάλλον προξενικών θεωρήσεων όπως ενεκρίθη από την Κομισιόν την 1η Απριλιά. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τεχνικού χαρακτήρα συναντήσεις ώστε να εξηγήσουμε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια όλες τις διαφορετικές πτυχές της προτάσης αυτής και φυσικά η διαδικασία αυτή θα ξεκινήσει η νομοθετική διαδικασία θα ξεκινήσει μόνο στο επόμενο κοινοβούλιο. Ευχαριστώ για την προσοχή σας κύριε Πρόεδρε και είμαι έτοιμο να απαντήσω σε τυχόν ερωτήματα σε αυτό το στάδιο. Ευχαριστώ. It's only obvious that... Uh, Είναι προφανές ότι για την Επιτροπή Λίμπη να διορίσει εισηγητές σε αυτά τα θέματα θα χρειαστεί πρώτα, ε, ε, ε, θα γίνει μετά τις εκλογές του Νέου Κοινοβουλίου, μετά το τέλος Μαΐου. Λοιπόν, Νομίζω ότι ο κύριος Μπρόγκ θέλει κάτι να πει. Ευχαριστώ καταρχήν την Επιτροπή που μας τα παρουσίασε. Ο κύριος Μπρόγκς, δεν θα με ακρηγορήσω. Στην αρχή της παρουσίας ακούσαμε ορισμένα στοιχεία ενδιαφέροντα που δείχνουν τα οικονομικά πλεονεκτήματα της διευκόλυνσης ή της απελευθέρωσης της χορήγηση θεωρήσεων. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ πιο εύκολο να υπολογίσει κανεί τα άτομα που επισκέπτονται τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αναρωτιέμαι πώ μπορούμε να υπολογίσουμε τα άτομα στα οποία δεν έχει χορηγηθεί θεώρηση, διότι αυτέ είναι οι δυσκολίε και αυτέ τι δυσκολίε θα έχουμε με τη διευκόλυνση χορηγήση θεωρήσεων. Είναι σαν να προσθέσουμε τους δύο πρώτους αριθμούς και μετά να τους υπολογίσουμε με δύο δεκαδικούς. Άλλα σχόλια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Εγώ θεωρώ ότι μπορούμε να αξιολογήσουμε θετικά το γεγονός ότι κινούμαστε προς λογικούς και ενιαίους κανόνες σε ό,τι αφορά τη χορήγηση προξενικών θεωρήσεων και θεωρώ επίσης θετικό ότι εκεί που βρίσκονται προβλήματα όπως παραδείγματος χάρη υπάρχει ιδιαίτερη πολυπλοκότητα και η υπερβολική γραφειοκρατία, υπάρχουν απαράδεκτες χρονικές προθεσμίες για την χορήγηση των θεωρήσεων, θα πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο. Και επίσης το να υπάρχει υποχρέωση εκπροσώπησης των χωρών που δεν έχουν ε, προξενικές αρχές. Έχουμε μια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, η οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και αυτή για να αντιμετωπίσουμε το θέμα των προξενικών θεωρήσεων δεν έχει νόημα να υποχρεώνουμε όλα τα κράτη-μέλη να έχουν προξενία όταν υπάρχει υπηρεσία εξωτερικής δράσης παρούσα. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και επίσης για μένα είναι θετικό το γεγονό ότι υπάρχει προβληματισμό για το να αντιμετωπίσουμε χωριστά αυτούς που είναι ερευνητές, ή επιχειρηματίες, ε, ταξιδιώτες, ή φοιτητέ κτλ. να έχουν τη δυνατότητα να έχουν μια προξενική θεώρηση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Όλα αυτά λοιπόν που έχουν να κάνουν με τη διευκόλυνση με βρίσκουν σύμφωνοι. Αλλά βλέπω και ορισμένα προβλήματα όπου νομίζω ότι η εκτίμηση της Κομισιόν αντίθετα από αυτά που είπε η Κομισιόν δεν είναι ε, οι καταλληλότεροι. Εγώ έχω άλλες αναφορές από τα κρατημέλη σε σχέση με τα προβλήματα αυτά. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα πρόβλημα στα σύνορα υπήρξε ένα πρόβλημα στα σύνορα της Βεντιμίλια μεταξύ Ιταλίας και Γαλλίας που αντιμετωπίσαμε προβλήματα στο παρελθόν γιατί είδαμε ότι η ευκολία με την οποία διηγόντουσαν οι προξενικέ θεωρίες θεωρήθηκε ως μια πηγή κατάχρησης και όλα αυτά οδήγησαν σε αντιπαραθέσεις μεταξύ Ιταλίας και Γαλλίας και ουσιαστικά αυτό οδήγησε και σε προβλήματα σε σχέση με, ε, με την κοινή αντιμετώπιση των προσφύγων διότι θεωρήθηκε ότι υπήρξε κατάχρηση του δικαιώματος για την ε, αίτηση ασύλου. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι αυτές οι αλλαγές που προτείνει η Κομισιόν είναι επαναστατικού χαρακτήρα. Εμένα με ενδιαφέρει να έχουν μεγαλύτερη ισορροπία. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη να έχουμε διευκολύνσεις αλλά και την ανάγκη να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια γιατί αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αφορά όλα τα κράτη-μέλη και είναι φανερό για μένα ότι δεν έχουν ληφθεί οι απαραίτητες διαφυλάξεις γιατί όταν ορισμένες κατηγορίες ε, δεν αντιμετωπίζουν, δεν αντιμετωπίζονται σωστά και υπάρχει αύξηση του κινδύνου πραγματικοί ταξιδιώτες να αντιμετωπίσουν προβλήματα. Πολλές φορές υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν επιτακτική ανάγκη να ταξιδεύσουν και θίγονται από αυτές τις ε, ε, λύσεις και είναι επίσης θέματα τα οποία πρέπει να έχουν μια ε, αντιμετώπιση από την Europol και Interpol όταν οι προξενικές θεωρήσεις οδηγούν σε καταχρήσεις και αυτό μπορεί να αφορά ακόμα και πολίτες της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γενικά φυσικά οι ταξιδιώτες Bonafide θα πρέπει να έχουν μια διευκόλυνση και εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ε, βράχυνση των, προξεν... της θεωρήσεων Ήδη σε πολλά κρατημέλη αυτό που λέμε οι 15 μέρες είναι πρόβλημα την περίοδο των Χριστουγέννων σε πολλά κρατημέλη γιατί είναι άφαντοι οι προξενικοί υπάλληλοι εκείνες τις μέρες και δεν μπορεί κανείς να πάρει τα έγγραφα αυτά. Εγώ νομίζω δεν πρέπει να αναφερόμαστε σε ημερολογιακές ημέρες στην προθεσμία αλλά σε εργάσιμες μέρες. Επίσης δεν αναφέρεται τίποτα για τις απαραίτητες χρηματοδοτήσεις την ε, ανάγκη να έχουν απαραίτητα ε, κονδύλια η καλή της πίστης, καλή πίστη ε, ταξιδιώτες. Εγώ δεν ξέρω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το Cirque du όπως αναφέρθηκε, αλλά ούτως ή άλλως δεν μπορεί αυτό να θεωρηθεί ότι είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εμείς θέλουμε να εξασφαλίσουμε τα θέματα ασφάλειας και γι' αυτό πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι ταξιδιώτες έχουν επαρκή χρήματα στα χέρια τους και για αυτό το θέμα νομίζω ότι θα πρέπει να παραμείνουμε στους κανόνες της προηγούμενης ρύθμισης, επομένως <clears throat> να πρέπει να αναλαμβάνουν την ε, υποχρέωση οι, ίδιοι οι ετούντες να αποδείξουν από τον τραπεζικό του λογαριασμό ότι έχουν τα απαραίτητα στοιχεία και όχι να είναι τα κράτη-μέλη τα οποία θα επομιστούν τον, το κόστος ενός ενδεχόμενου ταξιδιού επιστροφής. Είναι λοιπόν απαραίτητο να υπάρξει μια απόδειξη επαρκών οικονομικών δυνατοτήτων από τους ταξιδεύοντες και φυσικά και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν τις οικονομικές δυνατότητες γιατί αν το κάνουμε αυτό με τα κράτη-μέλη μπορούμε να, να προσκρούσουμε επομένως και σε προβλήματα προσωπικών δεδομένων. Θα πρέπει λοιπόν η ρύθμιση να γίνεται με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι λογικός και σε σχέση με τις βίζες πολλαπλού, πολλαπλής εισόδου τρία ή πέντε χρόνια νομίζω ότι αυτό έχει πραγματικά νόημα για φοιτητέ και θα πρέπει να προστατευτούν αυτοί από πολυπλοκότητα Ίσως θα υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιεί κανείς τα προηγούμενα έγγραφα που δόθη, με το βάση των οποίων δόθηκαν υποξενικές θεωρίες και να πιστοποιεί ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα και όχι να πρέπει να πάει κάποιος σε μια άλλη χώρα για να μπορέσει να αποκομίσει έγγραφα αυτά όταν υπάρχουν ε, δυσκολίες. Το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων όμως και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα και για τον ετούντα και το κράτος μέλος και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να εξασφαλίσουμε μια πιο εξισορροπημένη ε, λύση η οποία δεν θα οδηγήσει σε διαμάχες μεταξύ των κρατών μελών και θα αποκλείσει ορισμένα άτομα από την, από την δυνατότητα να κινηθούν θα πρέπει να εξασφαλίσουμε από τη μια μεριά τη δυνατότητα να μπορεί να κινείται κανεί μέσα σε εύλογα πλαίσια και από την άλλη μεριά να αντιμετωπίσουμε τι προφανείς απαιτήσει εξασφάλιση τη ασφάλεια που πρέπει να αντιμετωπιστεί από κάθε μέλη. Ευχαριστώ. Uh, ε, σχόλια από τα μέλη που βρίσκονται εδώ. Α επανέλθουμε στην Επιτροπή και κατόπιν ίσω η Ελληνική Προεδρία θέλει κάτι να προσθέσει. Ε, η Επιτροπή θέλει να αντιδράσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σχετικά με την πρώτη παρέμβαση που έγινε για τα στοιχεία των ταξιδιών που δεν έγιναν στο χώρο Σέγγεν, βεβαίως δεν έχουμε στοιχεία, έχουμε μόνο εκτιμήσεις αποτελέσματα μελετών που έχουν διενεργηθεί. Η Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων ε, παρήγγειλε μία μελέτη για τις οικονομικές επιπτώσεις ε, της ε, πολιτικής διευκόλυνσης των θεωρήσεων. Κατέληξαν λοιπόν με αυτά τα στοιχεία και παρόμοια στοιχεία έχουν κατατεθεί πέρσι μετά από τις συνεδριάσεις της, ε, ε, της Γενικής Διεύθυνσης Τουρισμού και των Υπουργών Τουρισμού που εξέτασαν τις επιπτώσεις από τη διευκόλυνση και την απελευθέρωση των θεωρήσεων. Πιστεύω ότι ε, δεν επιβεβαιώνονται τα στοιχεία αυτά οι εκτιμήσεις, αλλά νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουν αν κατέχει ένα άτομο μία θεώρηση με πολλαπλές εισόδους για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε αυτό το άτομο μπορεί να μεταβεί στις χώρες Σέγγεν ακόμα και για ένα Σαββατοκύριακο αυτά τα ταξίδια δεν θα γίνονταν εάν το άτομο αυτό θα πρέπει για ένα Σαββατοκύριακα να περάσει από όλη τη διαδικασία χορήγησης θεωρήσεων Σέγγεν. Βεβαίως οι εκτιμήσεις παραμένουν πάντοτε εκτιμήσεις, αλλά είναι σαφές ότι περισσότερα ταξίδια ε, στις χώρες Σέγγεν θα συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη αυτών των χωρών. Ε, κατόπιν το ίδιο άτομο έθεσε ορισμένα ερωτήματα, έκανε σχόλια που αφορούν σημαντικά θέματα, ε, τροπολογίες που προτείνει η Επιτροπή και πρέπει να συζητηθούν περαιτέρω. Θα ήθελα να κάνω λίγα σχόλια αυτή τη στιγμή. Το θέμα του βάρους που θα πρέπει να επομισθούν οι προξενικές αρχές των κρατών μελών. Οι προτάσεις που κατέθεσε η Επιτροπή δεν έχουν ως στόχο μόνο να διευκολύνουν ε, τη ζωή των νόμιμων ταξιδιωτών. Σκοπός μας είναι να βελτιώσουμε ε, την συνεργασία μεταξύ προξενικών αρχών και είναι βέβαιο ότι ορισμένα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή όπως τη πιο τακτική χορήγηση θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων με μεγάλη διάρκεια, θα ωφελήσουν ε, και θα μειώσουν το βάρος των προξενικών αρχών των κρατών μελών. Συνεπώς, αυτό δεν εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα του ετούντος, αλλά η πρόταση αυτή περιέχει στοιχεία που θα διευκολύνουν τη ζωή των προξενικών αρχών των κρατών μελών. Κατόπιν έγιναν σχόλια για το θέμα ε, της εμφάνισης του ατόμου που κάνει την αίτηση για θεώρηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο περιλαμβάνεται στον κώδικα περιθεωρήσεων. Αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη ότι ήδη 70% των ετούντων δεν εμφανίζονται αυτοπροσώπως στις προξενικές αρχές, αλλά πηγαίνουν σε ένα κατάστημα θεωρήσεων, το οποίο ε, διευθύνεται από έναν πάροχο εξωτερικών υπηρεσιών. Συνεπώς δεν υπάρχει άμεση επαφή μεταξύ του ετούντος και του προξενικού υπαλλήλου, ο οποίος θα χορηγήσει την θεώρηση. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, η εμφάνιση του ατόμου αυτοπροσώπως δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Αλλά η Επιτροπή εξακολουθεί να περιλαμβάνει στην πρόταση την υποχρέωση εμφάνιση αυτοπροσώπως την πρώτη φορά δηλαδή για το άτομο το οποίο δεν έχει καταγεγραμμένα τα στοιχεία του στα Μητρώα και στο VS, στο VIS. Από τη στιγμή που έχει καταγραφεί τότε υπάρχει ευελιξία σχετικά με την κατάθεση της αιτήσεώς του. Υπό αυτή την έννοια για ε, τον ε, υποχρέωση εμφάνιση από το προσώπο του ετούντου για πρώτη φορά εξακολουθεί να υπάρχει. Αυτό όμω δεν αφορά τι ε, μεταγενέστερε αιτήσει. Επίση, έχει ένα σχόλιο σχετικά με τι συνθήκε που τι οποίε παρέχεται αυτόματη χορήγηση θεωρήσεων με πολλαπλέ εισόδου με μεγάλη διάρκεια εγκυρότητα. Δεν υπάρχει απόλυτος αυτοματισμός. Η Επιτροπή πιστεύει ότι για τους ε, ταξιδιώτες που είναι εγγεγραμμένοι στο VIS, δηλαδή τα άτομα τα οποία έχουν ε, αποκτήσει ε, θεωρήσεις προηγουμένως και τις έχουν χρησιμοποιήσει σωστά, τότε αυτά τα άτομα υποφελούνται από την υπόθεση ότι διαθέτουν τα οικονομικά μέσα για να κάνουν το επόμενο ταξίδι τους. Και ότι επιθυμούν να κάνουν ε, ε, και άλλες επισκέψεις με αυτή την θεώρηση. Έχουμε δει ότι ορισμένα άτομα που έχουν κάνει δύο ταξίδια, ίσως και προηγούμενα, ε, την, τα προηγούμενα έτη στην περιοχή Σέγγεν, μπορούν να χρησιμοποιούν και νόμιμα θεμητά της, τη θεώρησή τους, χωρίς να δημιουργήσουν προβλήματα. Τώρα δεν θα πρέπει πάλι να περάσουν από όλη τη διαδικασία, να αποδείξουν ότι έχουν τα μέσα ε, να ε, επιβιώσουν στις χώρες που θα μεταβούν. Υπάρχει λοιπόν η υπόθεση ότι διαθέτουν τα μέσα με βάση την καλή χρήση της προηγούμενης θεώρησης. Αυτή η υπόθεση βεβαίως δεν είναι απόλυτη. Ε, μπορεί να αντιστραφεί. Εάν με, το, με τη σφραγίδα εισόδου και εξόδου στο διαβατήριο βλέπουμε ότι έμεινε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αυτό το άτομο, η προξενική αρχή μπορεί να μην του χορηγήσει μία θεώρηση με πολλαπλές εισόδους. Ε, αν θέλετε λοιπόν πολλά πρέπει να δούμε ακόμα και ίσως θα έπρεπε, ε, αλλά αναφέρουμε τώρα σε ε, τεχνικές λεπτομέρειες, θα πρέπει ίσως να εξηγήσουμε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο και τις συνέπειες των προτάσεων της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ντεκόιστερ. Τώρα ο κύριος Βούλγαρης για την Ελληνική Προεδρία. Thank you, Mr. Chairman. Good morning. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Οι προτάσεις αυτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι άκρο σημαντικές λόγω του συσχετισμού μεταξύ τη πολιτική των θεωρήσεων, τη σταθερότητα και τη ελευθερία κυκλοφορία καθώ και τη οικονομική ανάπτυξη. Η Προεδρία σκοπεύει αμέσω να ξεκινήσει την εξέταση και τι συζητήσει για την πρόταση στην αρμόδια ομάδα εργασία. Όμω την επόμενη εβδομάδα κιόλα έχουμε μια διήμερη συνεδρίαση 15 και 16 Απριλίου για τη συζήτηση του θέματο αυτού στην σχετική ομάδα και για, την υπόλοιπη, για το υπόλοιπο διάστημα της προεδρίας μας θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε το, το, το θέμα αυτό να προχωρήσει και να προωθηθεί όσο δυνατόν περισσότερο. Ευχαριστώ. Εκτός μικροφώνου ο Πρόεδρος. Και τώρα για τρεις προπαρασκευαστικές ε, εργασίες για τη μεταβατική περίοδο 2013 1 Δεκεμβρίου 2014 θα ακούσουμε μια παρουσίαση της νομικής υπηρεσίας και μετά θα ακούσουμε και τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου. Θα γνωρίζετε εδώ το ιστορικό του θέματος, πενταετής μεταβατική περίοδος για την ε, αναβολή της εφαρμογής των ε, Υπόθετων κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ποινικά και αστυνομικά ζητήματα πριν την 1η ε, Δεκεμβρίου 2014 και κυρίως ό,τι αφορά τη δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά το τέλος της μεταβατικής αυτής περίοδου, 1η ε, Δεκεμβρίου του 2014, το άρθρο 10 του πρωτοκόλου 36 των Ευρωπαϊκών Συνθήκων δίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο τη δυνατότητα να αποφασίσει το αργότερο ως 31 Μαΐου 2014 εάν θα συνεχίσει να εξαιρείται ή όχι από τα θέματα και τη συνεργασία ε, στην, στα αστυνομικά και ποινικά ζητήματα πριν, όπως ίσχυαν πριν την 1η Δεκεμβρίου 2009. Κατά συνέπεια, όλο το ε, κεκτημένο πρώην τρίτου πυλώνα που δεν έχει λισαβονοποιηθεί θα πάψει να ισχύει στον Ηνωμένο Βασίλειο από την 1η Δεκεμβρίου 2014. Με επιστολή ημερομηνία 24 Ιουλίου 2013, ο μόνιμο αντιπρόσωπο του Ηνωμένου Βασιλείου γνωστοποίησε στο Συμβούλιο του Ηνωμένου Βασίλειο, αποφάσισε να χρησιμοποιήσει την επιλογή αυτή, να την ασκήσει και να εξαιρεθεί από το κεκτημένο που ανήκε στον ε, πρώην τρίτο πυλώνα. Βάσει του πρωτοκόλλου 36, το Ηνωμένο Βασίλειο δύναται οποιαδήποτε στιγμή αργότερα να ε, κοινοποιήσει στο Συμβούλιο την επιθυμία του να επιστρέψει και να ξαναρχίσει να εφαρμόζει πράξεις που έπαψαν να ισχύουν βάσει της απόφασης εξαίρεσης. Ε, βάσει του άρθρου 10, εδάφιο 5 του πρωτοκόλλου 36, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επισήμως ανακοινώσει την πρόθεσή του να ξαναασκήσει και να εφαρμόσει 35 ε, νομοθετήματα που έχουν να κάνουν με το Εκτιμένο που αναφέραμε. Πέντε μέτρα που έχουν σχέση με το Σέγγεν και 30 που δεν ανήκουν στο, χώρο του Σέγγεν. Για να αποβευθεί το λειτουργικό και νομικό κενό, το Ηνωμένο Βασίλειο θα ήθελε η επίσημη ε, γνωστοποίηση για την επανεφαρμογή αυτών των 35 μέτρων και την έγκριση των σχετικών αποφάσεων που δίνουν τη δυνατότητα να ε, εφαρμοστούν την ίδια μέρα τα μέτρα να ισχύσουν από την 1η ε, Δεκεμβρίου του 2014 ημέρα Δευτέρα. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η κυβέρνησή του επιθυμούν να περατωθεί η εξέταση του καταλόγου των μέτρων προ επανεφαρμογή μέχρι τον Ιούνιο του 2014 και ζητούν πολιτική συμφωνία σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Συμβουλή μέχρι τον Ιούνιο 2014. Οι διαπραγματεύσει μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και τη αντιπροσωπείας του και ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Συμβούλιο ξεκίνησαν τον περασμένο μήνα. Ε, λόγω των ευρωεκλογών θα πρέπει να μπορέσει και το Κοινοβούλιο να εκφράσει την άποψή του σε σχέση με αυτό το σημαντικό ζήτημα. Το, η νομική υπηρεσία του Ευρωκοινοβουλίου θα παρουσιάσει το τι ισχύει για το θέμα αυτό βάσει του πρωτοκόλλου 36 των Ευρωπαϊκών Συνθηκών και μετά μπορούμε να έχουμε ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Προεδρία για αυτό το ε, κέριο σημασία ζήτημα για τον Ηνωμένο Βασίλειο. Το κατά πόσον δηλαδή τον Ηνωμένο Βασίλειο συμμετέχει ή όχι στο χώρο ελευθερίας δικαιοσύνης και ασφάλειας όπως διαμορφώνεται βάσει τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Α ακούσουμε τον κύριο Καγιόλα από την νομική υπηρεσία και μετά θα ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον εκπρόσωπό τη, από την Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνη και μετά την, τον εκπρόσωπο τη Ελληνική Προεδρία. Κύριε Καγιόλα. Σα ευχαριστώ. Σύντομο θα προσπαθήσω να είμαι. Αλλά επειδή πολύπλοκο το νομικό πλαίσιο, με την ε, άδειά σας θα χρησιμοποιήσω λίγο χρόνο με την εφαρμογή της συνθήκης του Λισαβόνα. Της Την 1η Δεκεμβρίου 2009 επήλθαν σημαντικές αλλαγές στις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μαζί με αυτές τις αλλαγές προβλέφθηκε ένα μεταβατικό καθεστώς για ένα από τα πρωτόκολλα τα οποία προσαρτούνται στην συνθήκη. Το πρωτόκολλο 36 για τις μεταβατικές προβλέψεις. Προβλέπει το πρωτόκολλο αυτό και προνοεί μεταξύ άλλων για μεταβατικές προβλέψεις σε σχέση με πράξεις που έχουν εγκριθεί πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009 στον τομέα της αστυνομικής και ιδιοκτικής συνεργασίας για τα ποινικά θέματα. Το άρθρο 10 του πρωτοκόλλου 36 θεσπίζει ένα μεταβατικό καθεστώς το οποίο θα εφαρμόζεται στις πράξεις οι οποίες έχουν εγκριθεί με βάση των προνοιών για συνεργασία διοκτικών αρχών, αστυνομικών και δικαστικών αρχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ήταν στον, πρώτο, στον πρώην τρίτο πυλώνα. Για, επομένως για αυτές τις πράξεις του τρίτου πυλώνα οι εξουσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του δικαστηρίου θα παραμείνουν όσοι είχαν πριν τεθεί σε εφαρμογή η συνθήκη της Λισαβόνας μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2014 εκτός αν τροποποιηθούν πριν από αυτή την ημερομηνία. Δηλαδή Μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή οι αρμοδιότητες της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα, περι, θα είναι περιορισμένες όπως ήταν την εποχή του πάλε ποτέ τρίτου πυλώνα. Το δικαστήριο θα μπορεί να δίνει μοναχά προδικαστικές αποφάσεις όταν ένα κράτος μέλος έχει κάνει μια δήλωση η οποία αποδέχεται την ε, δοσηδικία του δικαστηρίου. Σε περίπτωση τώρα άμεσων ενεργειών μόνο οι πράξεις, οι αγωγές για ακύρωση μπορούν να έλθουν στο δικαστήριο μόνο από ένα κράτος μέλος ή την Κομισιόν και μόνο εναντίον μιας απόφασης πλαισίου και μιας απόφασης, όχι όμως εναντίον όλων των πράξεων του τρίτου πυλώνα. Οι διαδικασίες επί παραβάση της Κομισιόν εναντίον ενός κράτους μέλους για μη εφαρμογή μιας πρώην του τρίτου πυλώνα πράξης δεν είναι πια καθόλου δυνατές. Επιπλέον, οι άμεσες δράσεις των πολιτών ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αποκλείονται μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2014. Μετά από αυτή την ημερομηνία, όλες οι πράξεις του παλιού τρίτου πυλώνα θα εξακολουθούν να ισχύουν, αλλά ως εάν είχαν εγκριθεί επί τη βάση των κανόνων της ε, Συνδίκης Λισαβόνας με πλήρες εξουσίες για την Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτοί οι κανόνες εφαρμόζονται καταρχήν σε όλα τα κράτη-μέλη, αλλά υπάρχουν ορισμένες ειδικέ πρόνοιες για τη Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Πρώτα, επειδή αυτές οι χώρες είτε αυτή τη στιγμή δεν μπορούν ή δεν υποχρεωμένες να συμμετέχουν σε πράξεις της ε, συνδίκης Λισαβόνα στον τομέα ελευθερία δικαιοσύνη και ασφάλεια, υπόκεινται σε ειδικό κανόνα σε σχέση με την τροποποίηση πράξεων του τρίτου πυλώνα από νέε νομοθετικέ πράξει. Εάν δεν μπουν στη διαδικασία του opt-in, η παλαιά πράξη του τρίτου πυλώνα θα εξακολουθεί να ισχύει για αυτές τις χώρες μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2014 και θα εφαρμόζεται και ο περιορισμός της εξουσίας του Δικαστηρίου και της Κομισιόν όπως ανέφερα προηγουμένως. Για όλες τις άλλες χώρες θα εφαρμόζεται το νέο καθεστώς της Λισαβόνας ακόμα και πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2014. Δεύτερον και πιο σημαντικότερότερο, λόγω του χρονικού πλαισίου, το άρθρο 10 του πρωτοκόλλου 36 επιτρέπει την λεγόμενη μαζική διαδικασία αυτοεξαίρεσης του Ηνωμένου Βασιλείου από όλες τις πράξεις του τρίτου πυλώνα που δεν θα έχουν τροποποιηθεί ε, πριν από την 1η 2014 ε, ή και μετά από αυτήν την ημερομηνία χωρίς αποτέλεσμα για το Ευρωπαϊκό για το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό το opt-out θα πρέπει να ασκηθεί μέχρι την 31η Μαΐου 2014 με κοινοποίηση του Ηνωμένου Βασιλείου προς το Συμβούλιο. Δεν προβλέπεται κανένας ε, ρόλος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτε καν ε, κοινοποίηση προς το Κοινοβούλιο που να προβλέπεται από τι συνθήκε. Εάν δώσει αυτή την κοινοποίηση το Ηνωμένο Βασίλειο, όλε οι πράξει του τρίτου πυλώνα, οι οποίε δεν έχουν τύχει τροποποίηση μετά τον Δεκέμβριο του 2009 ή που έχουν τροποποιηθεί μετά από αυτή την ημερομηνία αλλά δεν έχουν αποτέλεσμα για το Ηνωμένο Βασίλειο θα πάψουν να ισχύουν για το Ηνωμένο Βασίλειο από την 1η Δεκεμβρίου 2014 και το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ήδη στήσει μια τέτοια εξαίρεση το Δεκέμβριο του 2013. Το Συμβούλιο Δρόν, επί τη βάση μιας πρότασης της Κομισιόν, θα αποφασίσει για τις κατάλληλες μεταβατικές διατάξεις. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα συμμετάσχει στην έγκριση αυτής της απόφασης. Περαιτέρω, το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία προτάσει της Κομισιόν μπορεί να εγκρίνει μια απόφαση η οποία θα καθορίζει ότι το, Ευρωπαϊκό, το Ηνωμένο Βασίλειο θα φέρει το οικονομικό κόστος αυτών των αποφάσεων, εάν ληφθούν τέτοιες αποφάσεις, με τρόπο αδύρυτο ως αποτέλεσμα της παραχώρησης της δυνατότητας συμμετοχής τους στις πράξεις αυτές νομοθετικού χαρακτήρα. Δεν προβλέπεται και πάλι να παίξει κανένα ρόλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ηνωμένο Βασίλειο σε οποιαδήποτε στιγμή στη συνέχεια θα μπορέσει να κοινοποιήσει στο Συμβούλιο την θέλησή του να συμμετάσχει σε νομοθετικές πράξεις οι οποίες έχουν πάψει να ισχύουν για το Ηνωμένο Βασίλειο μετά από τη μαζική αυτοεξαίρεση. Opt-out στα ελληνικά. Αυτή η κοινοποίηση θα έχει το πολύπλοκο αποτέλεσμα ότι οι ρήτρε του πρωτοκόλου υπαριθμών 19 για το κεκτημένο του Σέγγεν ή του πρωτοκόλου για τη θέση της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου στο χώρο ε, τους ελευθερίας δικαιοσύνης και ασφάλειας, πρωτόκολλο 21, θα εφαρμόζονται. Για οποιαδήποτε πράξη λοιπόν η οποία βασίζεται στο κεκτημένο του Σέγγεν, το ΕΒ μπορεί να, τύχει, να ζητήσει να τύχει άδεια να συμμετάσχει σε συγκεκριμένα μέτρα του Σέγγεν επί τη βάση του ε, άρθρου 4 παράγραφος 1 αυτού του πρωτοκόλου. Αλλά δεν μπορεί να λάβει μέρος στο Ηνωμένο Βασίλειο σε μεμονωμένα μέτρα του Σέγγεν χωρίς να κάνει και πάλι opt-in στο συνολικό και συνεκτικό σώμα του κεκτημένου του Σέγγεν όπως αναφέρει και η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου υπόθεση C77 του 2005. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν και μια απόφαση του Συμβουλίου ομόφωνα με ψήφο και του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά όχι τη Ιρλανδία για το θέμα αυτό. Το Κοινοβούλιο δεν εμπλέκεται για όλε τι πράξει τρίτου πυλώνα που δεν είναι τμήμα του κεκτημένου του Σέγγεν. Η διαδικασία opt-in του, Ευρωπαϊ... του Ηνωμένου Βασιλείου θα είναι ουσιαστικά αυτόματη. Είτε η Κομισιόν θεωρεί λοιπόν ότι οι συνθήκε συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν εκπληρωθεί όπου η διαδικασία επανίστοχη στο opt-back-in, γίνεται πραγματικότητα με αποτελεσματικό τρόπο. Η Κομισιόν θα θεωρήσει ότι δεν έχουν εκπληρωθεί αυτές οι προποθέσει, οπότε θα θέσει μια καταληκτική ημερομηνία για το Ηνωμένο Βασίλειο για να κάνει τα απαραίτητα θεραπευτικά μέτρα. Εάν μετά από όλα αυτά το Συμβούλιο θεωρήσει ότι οι προποθέσει που έθεσε η Κομισιόν δεν έχουν εκπληρωθεί, μπορεί το θέμα αυτό να επανέλθει στο Συμβούλιο, το οποίο με ειδική πλειοψηφία των κρατών μελών θα αποφασίσει, των χωρών όπου εφαρμόσετε το μέτρο θα αποφασίσει. Το άρθρο 301, πρώτη παράγραφος μαζί με το άρθρο 16 παράγραφος 3 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ε, άρθρων, άρθρων 1 και 3 της ε, Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εφαρμοστούν. Είμαι κάπως ιδιαίτερα τεχνικός, αλλά όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για να σας δώσουμε το γενικό πλαίσιο για τη δυνατότητα το Ηνωμένο Βασίλειο να επανέλθει με opt-back in. Ούτω ή άλλω δεν μπορεί κανεί να εμποδίσει για πολιτικού λόγου το Ηνωμένο Βασίλειο από τη διαδικασία αυτή επανεισδοχή στο πιεκτημένο και το Κοινοβούλιο δεν έχει κανένα λόγο σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό το πολύπλοκο λοιπόν σύστημα προβλέπεται χωρί καμία κοινοβουλευτική εμπλοκή, αλλά αυτό είναι μια εξαίρεση στου γενικού κανόνε τη ε, συνθήκη βάσει των οποίων οι κανόνε τη Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά όργανα έχουν την ίδια εξουσία για τα θέματα αυτά και έναντι όλων των άλλων κρατών μελών. Μία εξαίρεση σε αυτού του κανόνε είναι η διαδικασία ενισχυμένη συνεργασία που θα πρέπει να χρησιμοποιείται ω τελική καταφυγή μέσα στα πλαίσια των μη αποκλειστικών αρμοδιοτήτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 9 κράτη-μέλη. Αλλά μια τέτοια συνεργασία θα μπορεί να ξεκινήσει από οποιοδήποτε κράτο μέλο σε οποιαδήποτε στιγμή βάσει του άρθρου 20 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το καθεστώ τώρα του της αυτοεξαίρεσης του Ηνωμένου Βασιλείου για τον χώρο ελευθερίας δικαιοσύνης και ασφάλειας ακολουθεί μια αντίθετη πορεία. Ο γενικό κανόνα εκεί είναι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει στην έγκριση μέτρων για τον χώρο ασφάλεια δικαιοσύνη κτλ. και δεν δεσμεύεται από αυτά. Αλλά έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει με οπτήν σε συγκεκριμένα μέτρα. Στο βαθμό των μέτρων που έχουν εγκριθεί πριν από τη συνθήκη τη Λισαβόνα, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει τη δυνατότητα μιας μαζικής αυτοεξαίρεσης opt-out και να επανέλθει βάση του άρθρου 10 του ε, πρωτοκόλλου 36. Σε αυτό το εξαιρετικά πολύπλοκο νομικό πλαίσιο τίθενται ορισμένα θέματα σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως λένε τα προήμια των πρωτοκόλλων 19 και 21. Για τα μελλοντικά κρατημέλη, οι συντάκτες της συνθήκης έχουν προτείνει, έχουν διαλέξει μια διαφορετική προσέγγιση τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το κεκτημένο του Σέγγεν. Το άρθρο 7 του πρωτοκόλλου 19 προβλέπει ότι για λόγους διαπραγματεύσεων για την εισδοχή νέων κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το κεκτημένο του Σέγγεν και άλλα συναφή μέτρα που έχουν εγκριθεί από τα δεσμικά όργανα μέσα στο πλαίσιο του Σέγγεν θα θεωρηθούν ω ένα κεκτημένο το οποίο πρέπει να γίνει αποδεκτό πλήρω από όλα τα κράτη-μέλη ή τι υποψήφιε για ένταξη χώρε. Προσπάθησα λοιπόν να σας δώσω τα βασικά στοιχεία σε σχέση με την εφαρμογή και τις συνέπειες του άρθρου 10 του πρωτοκόλλου 36. Φυσικά η νομική υπηρεσία είναι στη διάθεσή σας εάν έχετε ακόμα απορίες και χρειαζόσαστε πιο ενδελεχή μελέτη. Επιτροπή, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καθώς και την Επιτροπή Λίμπη που μας δίνει αυτή την ευκαιρία να σας εξηγήσουμε ποια είναι η κατάσταση σχετικά με το πρωτόκολλο 36 για τα μεταβατικά θέματα. Συμφωνώ με την Γενική Διεύθυνση Ιστονικών Υποθέσεων ότι αυτή είναι μια κοινή άσκηση και ευχαριστούμε πολύ επίσης τη νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτή την πολύ περιεκτική ανασκόπηση ε, του πρωτοκόλλου 36. Υπάρχουν δύο πλευρές στο πρωτόκολλο 36. Ε, το ένα έχει άμεση σχέση με το τέλος της μεταβατικής περίοδου και τις επιπτώσεις ε, από την υιοθέτηση ε, του, κεκτημένου, του επίσημου κεκτημένου του τρίτου πυλώνα στο τέλος περίοδου και το δεύτερο σκέλος έχει σχέση με το opt-out του Ηνωμένου Βασιλείου για το πρωτόκολλο 36. Αυτή τη στιγμή ασχολούμεθα με, τις τεχνικές, ε, με την τεχνική επεξεργασία και την προπαρασκευαστική εργασία. Όπως ε, εξηγήθηκε, έχουμε μία πενταετή μεταβατική περίοδο η οποία εκπνέει στο τέλος ε, του Νοεμβρίου 2014 και τότε συγκεκριμένα την 1η Δεκεμβρίου οι αρμοδιότητες Επιτροπής και του Δικαστηρίου θα ε, μεταφερθούν στο, στο κεκτημένο του τρίτου πυλώνα. Έχοντας αυτά υπόψη, η Επιτροπή πρόσφατα έστειλε ένα έγγραφο εργασίας στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο, το οποίο αναφέρει σε συντομία το ε, που βρίσκεται το κεκτημένο του τρίτου πυλώνα. Είναι ένα συνδυασμό θεμάτων εσωτερικών υποθέσεων και νομικών θεμάτων στο τομέα τη αστυνομική συνεργασία και τη νομική συνεργασία για τα ποινικά θέματα. Ο κατάλογος που έχουμε έχει ως αντικείμενο να βοηθήσει τα κράτη-μέλη σε συζητήσεις τους, να βοηθήσει συζήτηση για ε, το κεκτημένο του τρίτου πυλώνα και να διευκρινίσει θέματα σχετικά με το τι είναι ο κατάλογος για το μέλλον. Ο κατάλογος δεν είναι παρά προκαταρκτικός, δεν είναι οριστικός και δεν είναι δεσμευτικός. Μπορεί ακόμα να εξελιχθεί υπό το φως των νομοθετικών εξελίξεων όπως η οθέτηση μέτρων όπως γίνεται σήμερα αυτές τις μέρες και σε αυτή την περίπτωση αν υπάρχουν τροπολογίες ή άλλες αλλαγές θα πρέπει να ενημερώσουμε τον κατάλογο. Ο κατάλογος συζητείται αυτή τη στιγμή με τους εκπροσώπους των κρατών μελών του Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, αλλά και η Προεδρία έχει πολλά να πει. Στο τέλος της συζήτησης πιθανόν θα ενημερώσουμε το κατάλογο αυτό προκειμένου να παρουσιάζει σαφή εικόνα της κατάστασης και να δώσει στα κράτη-μέλη τα στοιχεία που χρειάζονται ε, για να προετοιμαστούν οι νέες αρμοδιότητες Επιτροπής ε, και ε, του Δικαστηρίου μετά από την 1η Δεκεμβρίου. Για το δεύτερο σκέλος τώρα. Για το opt-out του Ηνωμένου Βασιλείου εξηγήθηκε ότι το Ηνωμένο Βασιλείο χρησιμοποίησε την αρμοδιότητά του, την, την εξουσία του opt-out για τον τρίτο πυλώνα και ε, παρουσιάζει ένα κατάλογο 35 μέτρων συγκεκριμένα που αφορά τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις. Αυτή τη στιγμή γίνονται τεχνικές και νομικές συζητήσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τα μέτρα αυτά και θα αποφασίσει ένα το χρόνο η Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για το opt-in και αυτή τη στιγμή αναλύουμε, εξετάζουμε αυτά τα μέτρα υπό το φως των απαιτήσεων του πρωτοκόλου 36, όπως ορίζει το άρθρο 10 παράγραφος 5. Και το κείμενο αναφέρει ότι θα προσπαθήσουμε να, να εξασφαλίσουμε την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στους δύο αυτούς τομείς που θα επηρεάσουν τα πρακτικά θέματα και συμβόμενη πάντοτε τη συνοχή. Υπό το φως αυτών των θεμάτων ε, της ε, διαλειτουργικότητας και της συνοχής ε, εξετάζουμε την υπάρχουσα κατάσταση και τα θέματα που έχουν σχέση με το opt-in του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτά γίνονται αυτή τη στιγμή και συνεπώς δεν μπορούμε να επισέλθουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ουσία του θέματος. Αλλά Ελπίζω ότι σας έδωσα μια γενική εικόνα του πού βρισκόμαστε τώρα, πέραν ε, του νομικού πλαισίου που σας εξηγήθηκε, πού βρισκόμαστε από πλευράς Κομισιόν όσον αφορά την παρακολούθηση των τεχνικών και προπαρασκευαστικών εργασιών για το πρωτόκολλο 36. Τώρα μπορώ να δώσω το λόγο στον συνάδελφο από τη Γενική Διεύθυνση Ιστορικών Υποθέσεων. Thank you, Mr. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παρακαλώ. Όπως μόλις είπε η από το Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνη, παρακολουθούμε αυτή τη δικασία από κοινού με μεγάλη προσοχή, η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης και με τη συμμετοχή των νομικών μας υπηρεσιών. Με πολλές τεχνικές και νομικές ε, παρατηρήσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη και στα δύο σκέλη αυτού του ε, θέματος. Αυτό που αφορά τα κράτη-μέλη συνολικά και αυτά που αφορούν την εφαρμογή του πρωτοκόλλου σε ένα κράτος μέλος πρέπει να πω ότι η διαδικασία αυτή ευχαρίστως να παρουσιαστεί στο Κοινοβούλιο ε, για δίποτε στιγμή σας χρειαστεί κάποια περαιτέρω διευκρίνηση καθώς οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εργάζονται άκουπα για το θέμα αυτό. Ε, Προεδρία του Ελληνικού Συμβουλίου, ευχαριστώ. Πρόεδρε, σημαντικό και περίπλοκο ζήτημα. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ασκήσει το δικαίωμά του να εξαιρεθεί από το πρωτόκολλο 36 των συνθήκων και αυτό το δικαίωμα είναι πολύ σημαντικό. Η Προεδρία καταγράφει την πρόθεση του Ηνωμένου Βασιλείου σε κάποια μέτρα του δικαιοσύνη και εσωτερικών υποθέσεων από την 1η Δεκεμβρίου 2014 να έχει και πάλι συμμετοχή. Σε αυτό το πλαίσιο έχει συσταθεί μια ομάδα φίλων της Προεδρίας στο Συμβούλιο, ώστε να δούμε το κεκτημένο που ανήκει στον τρίτο πυλώνα και που θα αρχίσει να ισχύει για τα υπολοιπα κατεμελη κατεμέλια από 1η Δεκεμβρίου 2014. Στο πλαίσιο αυτό, η δυνατότητα συμπερίληψη του Ηνωμένου Βασιλείου έχει ήδη συζητηθεί. Στην ομάδα αυτή κοιτάζουμε τι ορίζει και το πρωτόκολλο 36 στο άρθρο 10 και εκεί λέγεται ότι τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο θα φροντίσουν να δημιουργήσουν την, το πλαίσιο ε, συμπερίληψη του Ηνωμένου Βασιλείου στα θέματα δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια ε, και ιστορικών υποθέσεων, μάλλον, όπω θα ζητηθεί. Το προ... Η Προεδρία θα φροντίσει να μην υπάρξουν εμπόδια στην ομαλή συμπερίληψη του Ρωμανού Βασιλείου. Ε, το Συμβούλιο θα είναι υπεύθυνο για τα μέτρα Σέγγεν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα μέτρα εκτό Σέγγεν. Απλώ από κοινού κοιτάζουμε τα θέματα αυτά, διότι είναι αλληλένδετα. Λόγω χάρη υπάρχουν εργαλεία που είναι ταυτόχρονα και στον χώρο του Σέγγεν και εκτό. Θα πρέπει λοιπόν αυτά να εξεταστούν προσεκτικά. Το έργο της ομάδας βρίσκεται στα προκαταρκτικά στάδια, έχουμε συναντηθεί δύο φορές και είναι πολύ νωρίς για να αντλήσουμε συμπεράσματα. Η επόμενη συνεδρίασή μας προβλέπεται την επόμενη Δευτέρα και Τρίτη και η Προεδρία ευχαρίστως να επανέλθει στην Επιτροπή σας για να παρουσιάσει τα πορίσματα της ε, συζήτησης στην ομάδα μας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Βούλγαρη. Τώρα υπάρχουν συνάδελφοι, κύριε Μπρόγκς. Ναι. Εξ όσων κατάλαβα, ένα από τα μέτρα που η Βρετανική κυβέρνηση λέει ότι θέλει να ασκήσει και να εφαρμόσει και πάλι είναι το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Άκουσα πολύ προσεκτικά τον εκπρόσωπο της νομικής υπηρεσίας Και δεν θα περάσω τώρα στο λαβύρινθο των προϋποθέσεων βάσει των οποίων μπορεί ή δεν μπορεί το Ηνωμένο Βασίλειο μεταγενέστερα να έχει opt-back in. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι η απόφαση να συμμετάσχει στο σύστημα του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης είναι ένα σοβαρότατο σφάλμα. Διότι το δικαστήριο στη χώρα εκτέλεσης δεν μπορεί να αρνηθεί την απέλαση βάσει ανεπαρκών αποδεκτικών στοιχείων ή έλλειψης αποδεκτικών στοιχείων. Μπορεί να αρνηθεί μόνο λόγω διαδικαστικού προβλήματος ή αναλογικότητας. Δεν είναι απλώς θέμα λοιπόν δικαιοδοσίας και ε, ε, εθνικής κυριαρχίας, αλλά είναι και θέμα δικαιοσύνης. Πρόεδρος, άλλα σχόλια. Κάποιος άλλος συνάδελφος θέλει να παρέμβει. για αυτήν την μοναδική ιδιαιτερότητα του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο πλαίσιο των όσων προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας. Όχι, δεν υπάρχουν άλλα σχόλια. Οπότε η συνέχεια της διαδικασίας είναι ότι τον Μάιο και τον Ιούνιο ε, η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα συνεχίσουν τις σχετικές συζητήσεις και η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ θα παρακολουθήσει το πώς εξελίχθηκαν μετά την επανεκλογή, μετά την εκλογή μάλλον του Νέου Κοινοβουλίου και αφού αρχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του. Περνάμε τώρα στο σημείο 10. Τροποποίηση του προπολογισμού για το γραφείο του Ευρωπαϊκού Συστήματος, της Συστήματος Στήριξης Ασύλου. ΕΑΣΟ. Σκοπός είναι να αρχίσει να συμμετέχει και η Ορδανία στο έργο της ε, ε, ε, α. καθώς και της Τινησίας και του Μαρόκου. Θα υπάρξει λοιπόν αλλαγή στον προπολογισμό του ΆΣΟ από το 2014 με ένα εκατομμύριο ευρώ επιπλέον με μία εν μέρη επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το πρόγραμμα 18 μηνών. Η ΆΣΟ έχει υποβάλει τα σχετικά έγγραφα και το Κοινοβούλιο σημειώνει την δράση της ΕΑΣΟ στην εξωτερική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βάσει της στρατηγικής για την εξωτερική μας πολιτική από τον, ε, Δεκέμβριο του 2013. Από τον του 2013. Καλωσορίζουμε εδώ τον κύριο Μάρκ Καμιλέρη, από το Γραφείο Στήριξη του Ευρωπαϊκού Ασύλου που θα μα δώσει περισσότερε πληροφορίε για το πρόγραμμα αυτό τη ΕΑΣΟ που καλύπτει την Ορδανία αλλά και την Frontex, το Μαρόκο και την Τινησία. Και μετά την παρουσίαση θα έχουμε συζήτηση. Κύριε Καμιλέρη, κύριε Καμιλέρη, εφόσον είστε εδώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως υπόθηκε και στο ενημερωτικό σημείωμα, εδώ Έχουμε την πρώτη δράση της ΕΑΣΟ στο, στην εξωτερική διάσταση του κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Αυτό το κονδύλι προκύπτει από ένα εργαλείο το εργαλείο της νομικής εταιρικής σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στα τέλη του 2012 διατέθηκε από την ΤΕΦΚΟ με 3,7 εκατομμύρια ώστε να ενθαρρυνθούν οι τρίτες χώρες να συμμετάσχουν στο έργο των ευρωπαϊκών οργανισμών. Η ΑΖΟ εξέφρασε το ενδιαφέρον της, υπέβαλε μια πρόταση συμμετοχής η οποία έγινε αποδεκτή, αλλά δεν είναι μόνη της εδώ η ΑΖΟ. Ε, είναι ένα κοινό ε, εγχείρημα με την Frontex, όμως βασικός ε, τον είναι το ΕΑΣΟ και κάποια από τα όσα προβλέπονται θα ε, δοθούν με υπεργολαβία στην Frontex, με τις σχετικές συμβατικές διευθυντήσεις που προβλέπονται πάντα. Οι δικαιούχοι είναι τρεις χώρες, όπως σωστά αναφέρεται, η Ορδανία, το Μαρόκο και η Τινησία. Δεν προβλέπονται προβλήματα στην, στο διακανονισμό με τον Μαρόκο και την, ε, την Ισία, όπου δεν θα υπάρχει και άμεση συμμετοχή ε, του ΕΑΣΟ, αλλά μόνο στη δράση με την Ιορδανία. Η απόφαση για τις τρεις αυτές χώρες και η επιλογή τους βασίστηκε στο ενδιαφέρον που εκδήλωσαν οι ίδιες, αλλά και στη σημασία που, έχει, που έχουν οι χώρες αυτές για το έργο των δύο οργανισμών. Οι τρεις αυτές χώρες είτε έχουν συνάψει, είτε έχουν διαπραγματευτεί, είτε πρόκειται να διαπραγματευτούν συμφωνία κινητικότητας με την Ευρωπαϊκή Ένωση που ήταν η βάση για τέτοιου είδους συνεργασία. Τα μέτρα που προβλέπονται σε αυτό το εγχείρημα είναι εισαγωγικά. Στόχος είναι να αρχίσουν να λειτουργούν εκεί οι οργανισμοί, οπότε κυρίως θα υπάρχει συζήτηση και αποστολή εμπειρογνωμών από τα κράτη-μέλη προ τι χώρε αυτέ μέσω τη ΕΑΣΟ και του Frontex έχει να κάνει με την ευθυγράμμιση του αργού ε, στι χώρε αυτέ, με παρατήρηση του τι κάνουν και αποστολή ανταλλαγή δηλαδή εμπειρογνωμόνων από τι χώρε αυτέ προ τα κράτη-μέλη, θεματικά σεμινάρια και εργαστήρια που θα οργανώνονται από την ΕΑΣΟ και τη Frontex για διαφορετικά θέματα προφανώ και μετάφραση σημαντικού υλικού, ύλης, ενώ για την ΕΑΣΟ θα μεταφραστούν τρία από τα 14 βασικά εγχειρίδια εκπαίδευσης που πραγματικά ήταν γνωστά ως κύκλος για το ευρωπαϊκό άσυλο. Αυτά είναι πολύ σημαντικά κείμενα για το χώρο του ασύλου διότι έχουν να κάνουν με τη διδασκαλία, ε, περιλαμβάνουν ένα σκέλος το οποίο διατίθεται στο διαδίκτυο και κάποιες ε, διαζώσεις ε, συνεδρίες. Με τη μέθοδο λοιπόν αυτή, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορέσουν μακροπρόθεσμα να γίνουν οι ίδιοι εκπαιδευτέ. Είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που πιστεύουμε ότι θα έχει πολλαπλασιαστικέ συνέπειε στι χώρε αυτέ. Και ένα μεγάλο μέρο τη προσπάθεια θα είναι να μεταφραστούν τα κερδία αυτά προ τα αραβικά, αλλά να διατεθούν και στο διαδίκτυο. Και βεβαίω αυτό αφορά τη μετάφραση και την ε, προσαρμογή των κειμένων που απαιτούνται συνολικότερα. Το ενακτήριο λάκτισμα θα το έχουμε στις 13 και 14 Μαΐου. Οι πρώτες επισκέψεις έχουν ήδη γίνει στην Ιορδανία και το Μαρόκο, από κοινού με τη Frontex, με την πλήρη συμμετοχή και στην προπαρασκευαστική φάση και στη μελλοντική με συμμετοχή των Γενικών Διευθύνσεων DEFCO και HOME. Και βεβαίω η αντιπροσωπή τη Ευρωπαϊκή Ένωση προς τι χώρε αυτέ, αλλά και η συνεργασία μα με τους υπόλοιπου ευρωπαϊκούς οργανισμούς ε, θα είναι συστηματική ώστε να μην υπάρχει επικάλυψη επανάληψη των προσπαθειών. Και τα κράτη-μέλη θα συμμετάσχουν στην ε, επιδίωξη των αποτελεσμάτων αυτού του εγχειρήματο και ήδη έχει εκφραστεί ενδιαφέρον από αρκετά κράτη-μέλη για να έχουν συμμετοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση κύριε Καμιλέρη. Σχόλια για το εγχείρημα αυτό της Άσο. Έχει κάποιος να σχολιάσει κάτι. Όχι. Νομίζω είμαστε πάρα πολύ γρήγοροι σήμερα. Έχουμε ξεπεράσει τις προβλέψεις μας. Ε, δεν είναι και περίεργο, είναι τέλος θητείας. Είναι χαμηλότερες οι προσδοκίες στην τελική ευθεία. Το επόμενο όμως σημείο είναι, έχει προβλεφθεί για τι 10.40. Και επειδή θα έχουμε έναν άλλο προσκεκλημένο μας από τη Γενική Διεθνή Δικαιοσύνη, θα έλεγα να γίνει ένα διάλειμμα. Ένα διάλειμμα και να επανέλθουμε σε μισή ώρα. Διάλειμμα για μισή ώρα λοιπόν. Θα ξαναρχίσουμε στις 10.40. Ευχαριστώ.